NDCR, ALDE, Πράσινη, EFDD και ENF, ορισμένε αιτήσει διορισμών και αλλαγή τη σύνθεση επιτροπών και αντιπροσωπιών. Οι εν λόγω τροποποιήσει θα συμπεριληφθούν στα πρακτικά τη σημερινή συνεδρίαση. Εφόσον δεν υποβληθούν παρατηρήσει έω την έγκριση των πρακτικών, οι εν λόγω διορισμοί θα θεωρηθούν ότι έχουν εγκριθεί. Να ενημερώσω επίση το Σώμα ότι μετά τη διακοπή της Συνόδου του Σεπτεμβρίου